όσον αφορά την ετοιμασία του νέου μέσου στα πλαίσια του νέου πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέντινγκ. Τελειώσαμε με το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση Wallis. Πρόκειται για πολιτικές για τη δέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Πάνω από μια δεκαετία τα συζητούμε. Ήρθε τώρα η ώρα να αναλυφθεί η δράση. Γιατί αυτό είναι η ώρα. Τώρα που χρειάζεται μια όθηση η αγορά. Και γι' αυτό και η νομική επιτροπή είναι υπέρ του. Υπάρχει ένα προαιρετικό μέσο. Άλλο. Δίκαιο συμβάσεων για φυσικά πρόσωπα αλλά και επιχειρήσει. Νομίζω αυτό θα βοηθούσε Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια σκληρά, αυστηρά κριτήρια τι το επόμενο βήμα. Θα πρέπει να έχουμε υψηλό επίπεδο προτασία του καταναλωτού. ή Υψηλότερο από ότι εις πολλά κρατημέλη. Να είναι εύκολο, φιλικό στον χρήστη και στις ΜΜΕ θα πρέπει να απονέμει παράσημα εις αυτούς οι οποίοι ασκούν εμπορία επί τη βάση αυτή, αυτού του αυτής της σύμβασης του προαιρετικού μέσου και αυτό θα πρέπει να γίνεται με τρόπο συμβατό με το εθνικό δίκαιο οπότε θα πρέπει να έχουμε ε, τα, στοιχεία τα οποία να βασίζονται σε αξιολόγηση επιπτώσεων να μπλέκεται το κοινοβούλιο και από αυτής της βάσης όπως προείπα τέρμα τα λόγια χρειάζεται τώρα να κάνουμε βήματα πρόοδου κάποιοι με νευρικότητα λένε γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε απλά την ιδέα της εργαλειοθήκης. Εγώ εις αυτούς έχω να απαντήσω. Προσέξτε πολύ. Διότι διατηρώ κάποιες υποψίες ότι η εργαλειοθήκη χωρίς το προαιρετικό μέσο ενδεχομένως είναι ακόμα χειρότερη και ρίχνει το εθνικό δίκαιο από ότι το η εργαλειοθήκη με το προαιρετικό μέσο το οποίο χρησιμοποιείται κουσίω τα συμβαλόμενα μέρη τα σέβεται, τη βούλησή του, δηλαδή και είναι συμβατό με το εθνικό δίκαιο οπότε α κάνουμε το βήμα προόδου με αυτόν τον τρόπο και, έτσι να έχουμε προληπτική παρέμβαση τη δικαιοσύνη και έτσι να έχουν όλοι νομικά και φυσικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι το οποίο να του οδηγεί με δικαιοσύνη ή στην ανάπτυξη τέρμα τα λόγια, α κάνουμε βήματα προόδου. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινούμε τη διαδικασία Catch the Eye. είναι ο πρώτος συνάδελφος που θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Επίτροπε, συγχαίρω την κυρία Βόλη για τη δουλειά που έκανε και για το περιεχόμενο τη έκθεση τη, ε, την οποία υποστηρίζω πλήρω. Πιστεύω μάλιστα ότι μόνο αυτό το προαιρετικό μέσο που θα πενθετηθεί τη μέσω κανονισμού μπορεί τελικά να πετύχει του στόχου όλη τη μεταρρύθμιση όσον αφορά το δίκαιο των Ευρωπαϊκών Συμβάσεων. Ένα μέσο λοιπόν προαιρετικό δεν θα εναρμονίσει ούτε θα αντικαταστήσει το συμβατικό δίκαιο των κρατών μέλων. Αντίθετα, θα συνοδεύει αυτά τα μέτρα προσφέροντας ένα εναλλακτικό μέσο και ελεύθερη επιλογή για τα συμβαλόμενα μέρη. Δεν συμμερίζομαι λοιπόν τις προτάσεις που έκαναν εκείνοι που θέλουν να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής αυτού του μέσου μόνο στις συμβάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό δημιουργούσε μια διαφοροποίηση τεχνητή και πάνω απ' όλα άχρηστη μεταξύ online συναλλαγών και άμεσων συναλλαγών. Δική μας αρμοδιότητα δεν είναι να εξαλείψουν νομική φύση του κανονισμού ε, λόγω ε, κερδοσκοπιών της αγοράς, αλλά σαν νομοθέτες θέλουμε να εγγυθούμε ασφάλεια δικαίου και να θέσουμε τη βάση για μια κοινή νομική γλώσσα όσον αφορά τα εμπορικά ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαλτασάρη. Η κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρία Ρέντινγκ. Νομίζω το συμβατικό δίκαιο της Ευρώπης λειτουργεί με έναν τρόπο που στο τέλος θα πρέπει να αποφέρει θετικά αποτελέσματα κυρίως στους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί σήμερα βλέπουμε ότι οι πιο αδύναμοι των συμβαλόμενων μερών, δηλαδή οι καταναλωτές, χρειάζονται σήμερα στήριξη. Η κυρία Βόλης προτείνει αυτό το προαιρετικό μέσο έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν περισσότερα κίνητρα και ενθαρρύνσεις οι Ευρωπαίοι πολίτες. Οι καταναλωτές στην Ευρώπη θα πρέπει να βρουν τρόπο να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι ευρωπαϊκές συμβάσεις και να στηρίξουν τη θέση τους έναντι των επιχειρήσεων. Αυτό το προαιρετικό μέσο Βεβαίως αποτελεί μια προστασία, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και όλες τις άλλες δυνατότητες που εμπεριέχει αυτή η εργαλειοθήκη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέγνερ. Ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Wallace Πολύ γενναίο το βήμα που κάνει. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί η πρωτοβουλία, αλλά σίγουρα πρέπει να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε την όλη κατάσταση. Να την κάνουν πιο δίκαιη για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Να μπορούν οι καταναλωτές να αγοράζουν με τον ίδιο τρόπο στην πατρίδα τους και στο εξωτερικό. Όσον αφορά τις επιπλοκές που δημιουργούνται από την εθνική νομοθεσία. Ένα προαιρετικό μέσο, ένα σύστημα που μπορεί με προαιρετικό τρόπο να ισχύσει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, όμως πιθανότατα δεν είναι βιώσιμη. Πιθανότατα θα αντιμετωπίσει πολλά διαφορετικά νομικά συστήματα και εκεί θα κολλήσει, αλλά αξίζει τον κόπο η προσπάθεια. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα άλλωστε. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνοντα την ε, διαδικασία, Κατσδιάη ή η κυρια Ρόιτοβα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αυτό το προαιρετικό μέσο για τις συμβάσεις έχει ελαττώματα, αλλά και είναι ένας τρόπος εξαλείψεως των διαφορών όσον αφορά το συμβασιακό δίκαιο, που οδηγεί σε ποσοστό αποτυχίας 60% όσον αφορά τις διασυνοριακές παραγγελίες για τους καταναλωτές θα βοηθήσει και τι εταιρείε όσον αφορά το συμβασιακό νόμο, το νόμο για του καταναλωτέ, λογιστικέ προδιαγραφέ κλπ. κλπ. Σε 10 χώρε οι καταναλωτέ δεν μπορούσαν να, να βρουν πάνω από 50% από τα 100 προϊόντα που ήταν στις δοκιμές και μπορούσαν να τα βρουν πιο φθηνά σε άλλες χώρες. Γι' αυτό χρειάζονται τυποποιημένε συμβάσει μεταφρασμένε όλε τι γλώσσε για να διευκολυνθούν οι καταναλωτέ. Πρέπει όμω να αντιμετωπιστούν πάρα πολλά προβλήματα σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρόιτοβα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ΚΑΤΔΙ. Θα δώσω αμέσω το λόγο στην Επίτροπο, Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή, κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Wallis αλλά και τον κύριο Μάγερ και Πέτη Κάνεν για την εξαιρετική τους εργασία. Είναι σαφές ότι σήμερα βρισκόμαστε εν ώψη μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα και να προωθήσουμε την εσωτερική αγορά. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη, θέσεις απασχόλησης και καινοτομία. Πώς έχει όμως η κατάσταση μία στις τέσσερις επιχειρήσεις έχουν διασυνοριακές συναλλαγές μόνο. Και το εμπόριο αυτό περιορίζεται σε κάποια μόνο κράτη μέλη. Άρα δεν χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες που προσφέρει η εσωτερική αγορά. Οι καταναλωτές δεν μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά με αυτόν τον τρόπο, διότι οι παραγγελίες, οι διασυνοριακές, ξεπερνούν το 61%, μάλλον το 61% των ε, παραγγελιών αυτών εκτός των συνόρων δεν ολοκληρώνονται, αποτυγχάνουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η εσωτερική αγορά δεν αποφέρει τα ωφέλη που θα έπρεπε ούτε για τους καταναλωτές ούτε για τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ε, γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είδαμε ότι οι αποτυχίες, οι αδυναμίες της εσωτερικής αγοράς εν μέρη οφείλονται στις διαφορές μεταξύ των ε, νομοθεσιών των κρατών μελών. Πρόσφατα, μια έρευνα του Ευρωμαρόδου έδειξε ότι πραγματικά υπάρχουν 11 εμπόδια για αυτές τις εμπορικές συναλλαγές εμπόδια μεταξύ του καταναλωτή και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και να εξαλείψουμε μία προς μία αυτές τις δυσκολίες και αυτά τα εμπόδια. Γι' αυτό και η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια εδώ στο Κοινοβούλιο έχει, πρέπει να σας πω, ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια εκτός του Κοινοβουλίου. Έχει γίνει λοιπόν τεράστια προσπάθεια ανάλυσης. Οι προτάσεις έχουν υποβληθεί και γι' αυτό και συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι ήρθε η ώρα να δράσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Σημείωσα τις προτάσεις της ε, έκθεσης που αφορούν την πράσινη βίβλο, την στήριξη των ε, λύσεων που προτείνουν καινοτομία, που δεν στηρίζουν την εναρμόνιση αλλά που δίνουν ευκαιρίες στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν ένα ευρωπαϊκό ενιαίο σύστημα. Επίσης άκουσα ότι στηρίζεται ένα μέσο που θα μπορεί να λειτουργήσει στις συναλλαγές B2B και B2C. Δηλαδή συμβάσεις πωλήσεων, συμβάσεις για ψηφιακό περιεχόμενο, αλλά και προσφορά υπηρεσιών. Σημείωσα επίσης αυτά που είπατε ότι κάθε μελλοντικό μέσο, όποιο και να είναι αυτό, όποια και να είναι η μορφή του, θα πρέπει να προστατεύουν τον καταναλωτή έτσι ώστε να μην αποδυναμώσουν την προστασία του εθνικού δικαίου. Αλλά αυτό είναι μια προϋπόθεση. Εάν δεν πετύχουμε αυτή την προστασία θα αποτύχουμε στις προσπαθίες μας. Στις 3 Μαΐου η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας των ε, εμπειρογνωμόνων στο Συμβατικό Δίκαιο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητήσαμε από όλα τα συμβαλώμανα μέρη να σχολιάσουν και αυτή τη στιγμή η Επιτροπή αναλύει τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης και γίνεται και αξιολόγηση αντικτύπου έτσι ώστε να δούμε ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα με σκοπό να δώσουμε ένα κίνητρο στην εσωτερική αγορά σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσης, να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, θέσεις απασχόλησης να επεκτείνουμε την αγορά και να δώσουμε δυνατότητες για καλύτερη επιλογή, για καλύτερες συναλλαγές στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέντινγκ. Ολοκληρώσαμε και το θέμα αυτό. Αύριο στις 12 θα γίνει η ψηφοφορία. Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση Hirsch.